An excellent good morning to all of you. We... Καλημέρα σας. Περιμένουμε ήδη ένα-δυο λεπτά. Ξέρουμε ότι είναι 5 Δεκεμβρίου, είναι και 5η. Αλλά τώρα θα ξεκινάσουμε την κοινή μα συνεδρίαση, ΦΑΜ για σήμερα το πρωί. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω θερμό τον κύριο Τομπέ, τον πρόεδρο της Επιτροπής ΔΕΒΕ και βεβαίως όλα τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ, της Επιτροπής ΘΑΜ που είναι προσκεκλημένοι όλοι και προσκεκλημένες όλοι εδώ. Ε, η κοινή μα ατζέντα προβλέπει την 25η επέτειο τη Διεθνού Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, ICPD 25, την λεγόμενη Σύνοδο του Ναρόμπι. Και ε, θα μιλήσουμε και για την επίσκεψη εκεί την, των Επιτροπών ΘΑΜ και ΔΕΒΕ. Έχουμε λοιπόν τα δύο σημεία ταυτόχρονα τις ε, τροπολογίες, το ψήφισμα, τα πάντα και την ε, έκθεση προφανώς. Ε, πριν ξεκινήσουμε για να πάρουμε μέρος στην διάσκεψη ICPD 25 του Ναϊρόμπι, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΦΑΜ είχε μια ανταλλαγή απόψεων στις 6 Νοεμβρίου για το σχέδιο ψηφίσματος και μόλι επιστρέψαμε από τη Συνοδό, υπήρχε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στι 26 Νοεμβρίου. Έλεγε στι 26 Νοεμβρίου. Το πήραμε πολύ σοβαρά στην Επιτροπή ΦΑΜ και από ό,τι φαίνεται υποβλήθηκαν 209 τροπολογίε. Αυτό είναι το βασικό θέμα και αυτέ θα συζητήσουμε σήμερα. Επιπλέον, όπω ξέρετε, το σχέδιο προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχει κυκλοφορήσει για του χιώδει συζητητέ και αναμένουμε τι δικέ σα αντιδράσει. Τώρα, ως συνεισηγητή ε, για το θέμα αυτό, ε, θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο για μια σύντομη επισκόπηση για όλες αυτές τις τροπολογίες. Είναι πάρα πολλές, από ό,τι φαίνεται όλοι είναι πολύ ταγμένοι από το σκοπό. θα δώσω το λόγο στον συνεισηγητή και θα ήθελα να πω ότι αυτό που φαίνεται από τις τροπολογίες είναι ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά δεδομένα. Ε, πρέπει να βασιζόμαστε σε στοιχεία και δεδομένα για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα για το... Ε, για την εξέλιξη του πληθυσμού το 2018 και να έχουμε μια συνολική εικόνα ε, για την κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στον κόσμο σήμερα. Επιπλέον, πρέπει να ενισχύσουμε το σχέδιο ψηφίσματος με επιπλέον αναφορές στους αναπτυξιακού στόχους και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά είναι ε, ξεκάθαρα νομίζω και επίσης να είναι σαφής ο συσχετισμός μεταξύ της υλοποίησης και της πραγματικής άσκησης δικαιωμάτων σεξουαλικής αναπαραγωγικής ε, υγείας για γυναίκες και κορίτσια. Επίσης πρέπει να έχουμε, με συγχωρείτε τα αγγλικά μου είναι λίγο μαγκωμένα το πρωί, ε, πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένες αναφορές στον ακριτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων και τους καταναγκαστικούς γάμους για παιδιά και επίση όλα τα δικαιώματα σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, όπω την πρόσβαση σε υγειονομική, ε, περίθαλψη ή αγωγή. Γιατί ιδάλω μπορεί να υπάρχει κάποια μορφή έμφυλη βία, άσκηση βία κατά των γυναικών και κοριτσιών φυσικά. Εδώ σημαντικό είναι να εγκριθεί και η ε, σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονίσουμε ε, τι ευπρόσδεκτε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο, ώστε να αποδώσει 29 εκατομμύρια ευρώ για τα θέματα αυτά και να τονίσουμε ότι το καθολικό πακέτο των υπηρεσιών σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία θα πρέπει να καλύπτουν και αυτέ τι υπηρεσίε που ως τώρα δεν έχουν χρηματοδοτηθεί αρκετά. Όπω την αγωγή κατά της στηρότητας, την ε, ε, θεραπεία από πράξεις σεξουαλικής βίας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το αντικείμενο των περισσότερων τροπολογιών που έχουν υποβληθεί ως τώρα και με αυτά τα λόγια θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συμπρόεδρό μας, τον κύριο Τομπέ. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλες και όλους. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω πόσο σημαντικό θεωρώ ότι μπορούν να συνεργαστούν οι δυο μας επιτροπές για τα θέματα αυτά. Ιδίως για τα θέματα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να δούμε τι ευκαιρίε έχουμε για να αναπτύξουμε νέε μορφέ συνεργασία μεταξύ μα. Το σχέδιο ψηφίσματο, κατά την άποψή μου, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και καλά κάνουμε και οργανώνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα, όπω είχαμε κάνει και μετά την Σύνοδο. Το κοινό ψήφισμα σκοπό έχει να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα ως προς την επιταχυμένη εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ιδίως του ε, οικειοθελούς ε, οικογενειακού σχεδιασμού, της χειραφέτησης των γυναικών και της καταπολέμησης της εμφυλής βίας. Εάν θέλουμε να ολοκληρώσουμε όσα δεν έχουν γίνει ακόμα μετά την σύνοδο ICPD που είχε γίνει πριν από 25 χρόνια, την πρώτη, ε, θα δούμε ότι η τωρινή η σύνοδος του Ναρόμπι ήταν μια μεγάλη επιτυχία με 9.000 συμμετοχές, με νέες ενώσεις και κυβερνητικούς εκπροσώπους, μη ε, κυβερνητικές ε, οργανώσεις, ε, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ό,τι καθεξής. Έτσι καταλήξαμε στη δήλωση του Ναϊρόμπι για τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας περιθμών 25 με πολλά καλά αποτελέσματα. Θέλω να τονίσω ότι όλοι οι βουλευτές εργάστηκαν επικοδομητικά κατά τη διάρκεια της Συνόδου και στις συνεντεύξεις τύπου που διοργανώθηκαν μετά. Είναι δική μας λοιπόν ευθύνη τώρα να ελέγξουμε την πρόοδο και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στην Επιτροπή Ανάπτυξη θα παρακολουθούμε εάν τηρούνται οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί και από την Επιτροπό μα, την κυρία Γιουπλάινεν και όπως είπε η συμπρόεδρος έχουμε λάβει μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Να δηλώσω ότι προσωπικώς είμαι έτοιμη, έτοιμος να ενισχύσω αυτές που θα τονίσουν τις μνήες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπερμάχου των οικονομικών μας δεσμεύσεων για τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να δούμε και τα σχετικά εργαλεία αναπτυξιακή βοήθεια και στο πλαίσιο του ε, επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να τονίσουμε και το ρόλο τη κοινωνία των πολιτών και των ε, μεκυβερνητικών κυβερνητικών οργανώσεων για το πρόγραμμα δράση ε, για τα για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και την εφαρμογή του. Τι επόμενε εβδομάδε θα προτείνουμε μια σειρά από συμβαστικέ προτάσει ω συνεισηγητέ και να τονίσω ότι θεωρώ σημαντικό να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συγκλίνουν οι απόψει μα. Διότι αυτό είναι το βασικό, ότι πρέπει να συγκλίνουμε κάπω για να βρούμε τι καλύτερε δυνατέ συμβαστικέ λύσει. Ε, με αυτά και με αυτά, να δώσω το λόγο στους κοιόδους εισηγητές των Επιτροπών Ντέβε και ΦΑΜ να πάρουν το λόγο. Πρώτα απ' όλα ο λόγος στην κυρία Φιτζέραλτ από το ΕΛΚ. Thank you very um, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω οι δύο επιτροπές, τις δύο επιτροπές που συνδύασαν αυτήν την ακροασή. Αν είχε κανείς πια αμφιβολία γι' αυτό, το Ναϊρόμπι έδειξε ότι οπωσδήποτε πρέπει να συνεργαστούμε λόγω των θεμάτων που έφυγησαν και Θέλω να συγχαρώ την ηγεσία της αντιπροσωπείας. Πιστεύω πως δουλέψαμε αποτελεσματικά όσον αφορά την ε, διάδοση και την γνωστοποίηση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε και στο μέλλον ότι η εργασία μας και ο ρόλος μας θα εντάσσεται ακόμη περισσότερο στα προγράμματα. Ζητήσαμε από τις γραμματείες των δύο επιτροπών να το εξετάσουν αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα διάφορες σημαντικές διασκέψεις του ΟΗΕ ε, που είναι προγραμματισμένες. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να μην ε, χωριστούμε και να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, εφόσον δηλαδή υποδείξουμε αρκετά νωρίς ότι θα συμμετέχουμε, να μην κάνουμε μετά πίσω. Δεύτερον, η συμμετοχή των νέων στη διάσκεψη με ευχαρίστησε ε, ειδικά νέοι άνδρες που συμμετείχαν και ε, ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Φυσικά και θα πρέπει περισσότεροι να συμμετέχουν. Όμως η κλίμακα των ζητημάτων που προέκυψαν από αυτή την διάσκεψη, όπως πρόσβαση στην αντισύλληψη, ε, ήταν τρομακτική. Περισσότεροι γνωρίζαμε την κλίμακα πριν πάμε. Έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα και θέλω να στηρίξω τα όσα είπατε για την επιτάχυνση της ενημέρωσης ε, και ε, να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε με σοβαρό τρόπο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και να προσέξουμε όσο μπορούμε περισσότερο, διότι οι ανάγκε είναι τεράστιε. Μπορούμε να παίξουμε θετικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου. Τρίτη παρατήρηση ήταν κάτι που με απογοήτευσε πάρα πολύ. Ήταν η αμερικανική προσέγγιση στη διάσκεψη και αυτό πρέπει να ε, το ονοματίσουμε με την έννοια ότι οι Αμερικανοί, ο Αμερικανό πρέσβη έκανε έκανε άλλη συνέντευξη τύπου, έκανε εναλλακτικέ συζητήσεις και υπήρξαν διάφοροι που θέλησαν να υποβαθμίσουν, να υπονομεύσουν τη διάσκεψη. Αλλά αυτό ήταν, ε, είχαμε καταπληκτική επαφή με τον Διευθυντή στη διάρκεια της ε, διάσκεψης μας είπε πως πολύ περισσότεροι ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διάσκεψη, χιλιάδες που ήθελαν να παρακολουθήσουν αλλά δεν μπόρεσαν για πρακτικούς λόγους. Πρέπει λοιπόν να γιορτάσουμε αυτήν την διάσκεψη γιατί στηρίχθηκε από τη διεθνή κοινότητα και σας ευχαριστώ άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Uh, just want σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την διάσκεψη και την συνέντευξη τύπου που κάναμε από κοινού οι Επιτροπές ΦΑΜ και ΝΤΕΒΕ στο Ναϊρόμπι. Όπως μόλις ακούσαμε, όλοι απογοητευτήκαμε από την, το τελικό αποτέλεσμα γιατί ε, τελικά γύρω στις 20 χώρες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ε, ήταν ε, η θέση του επίμαχη σε σχέση με τα πορίσματα της διάσκεψης ανάμεσα στις χώρες αυτές ήταν σημαντικές νομίζω χώρες της Αφρικής αλλά και δύο ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, Πολωνία και Ουγγαρία. Όταν κάναμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου αυτό το τονίσαμε ότι δεν είμαστε δηλαδή σε θέση να μιλήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με μια φωνή. Το συμπέρασμα όμως είναι ότι για μένα ε, είναι ότι θα πρέπει να συζητήσουμε για το τι γίνεται με αυτά τα δύο κράτη-μέλη. Νομίζω πως ε, δεν είναι καλό το να ε, ε, κατηγορήσουμε και να τιμωρήσουμε αυτές τις δύο χώρες. Έχουμε τα καλύτερα μέσα όσον αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό, την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θα πρέπει λοιπόν καλύτερα να έρθουμε σε συζήτηση με την Πολωνία και την Ουγγαρία για να μας εξηγήσουν, αυτοί οφείλουν να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν μπόρεσαν να συμβαδίσουν και πιστεύω πως υπάρχουν δυνατότητες να τους πείσουμε διότι τόσα πολλά μέλη του ΦΙΝΤΕΣ για παράδειγμα και του ECR που είναι πολύ κοντά στις απόψεις μας όσον αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αυτή είναι η δική μου πρόταση, ότι δηλαδή θα πρέπει να, ε, να φεύγουμε μια νέα στρατηγική και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τα δύο κράτη-μέλη που διαφωνούν μαζί μας. Να ευχαριστήσω όμως την αντιπροσωπεία στην Ρέμπη που έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά ε, ειδικά όταν προέκυψε σύγκρουση για τον χρονισμό της διάσκεψης ε, της ε, συνάντευξης τύπου τον είπα και τη δική μας και για να τα πω ανοιχτά νομίζω πως επιτύχαμε γιατί Τελικά ήμασταν λίγο πιο πονηροί από τους Αμερικανούς. Ήταν όμως απαραίτητο να πετύχουμε. Και είχαμε μια καλή συνέντευξη τύπου όλα τα μέσα της ε, <coughs> μαζικής ενημέρωσης της Κένια ήταν παρόντα και δεν ήταν εύκολο να τους πείσουμε για τις δικές μας απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, ήταν πολύ θετικό που συζητάμε για αυτό το κοινοψήφισμα. Ε, και είναι πραγματικά δύνατο να μην το συζητήσουμε, αλλά να σας πω ότι θα γίνει και άλλη συζήτηση όταν θα χρειαστεί ε, με τις χώρες αυτές. Αυτά λοιπόν, να δώσω το λόγο στην κυρία Ζαχαροπούλου. Καλημέρα σας. Θα τα πω θα, αρχικά στα αγγλικά και μετά θα μιλήσω γαλλικά. Καταρχάς, αγαπητή Εύελιν και αγαπητέ Τωμά, ε, σε, ευχαριστώ πολύ, διότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε αυτή τη συνεργασία μεταξύ των Επιτροπών ΦΑΜ και ΝΤΕΒΕ και αυτό το πνεύμα το ομαδικό στη διάρκεια αυτής της αποστολής. Πιστεύω <clears throat> ότι αυτός ο συνδυασμός γυναικών και επιτροπών γυναικών και επιτροπών ανάπτυξης, επιτροπής ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί μαζί μπορούμε να μεταφέρουμε ε, την ευρωπαϊκή φωνή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα γυναικεία δικαιώματα εκτός Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες και τώρα θα μιλήσω γαλλικά. Ε, στο όνομα της ομάδας Renew προτείνουμε 26 τροπολογίες με στόχο να ενισχύσουμε το κείμενο του ψηφίσματος κυρίως για τα εξή στοιχεία. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το πνεύμα του Ναϊρόμπι και να το εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που στόχο θα έχει την αυτονόμηση των γυναικών και των κοριτσιών και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Να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 η ΟΗΕ θα διοργανώσει στο Μεξικό και στο Παρίσι το 2020 και θα γιορτάσει την επέτειο της δήλωσης του Πεκίνου το 2020. Τα δικαιώματα των γυναικών, η υποχώρηση των δικαιωμάτων των γυναικών και κυρίως του δικαιώματος ε, αυτοδιάθεσης του σώματός τους παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στην Ευρώπη. Σημαντικό είναι να υπάρχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ε, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα. Επίσης, η πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, η στρατηγική ε, καταπολέμησης του ε, ιού του HIV και κυρίως στην, ε, στην Ποσαχάρη Αφρική, είδαμε την ανάγκη επίσης να ε, συμπεριληφθεί μια ολόκληρη σειρά ανθρώπων από ανθρωπιστική άποψη ώστε να προστατευτούν καλύτερα από τη βία στην οποία είναι εκτεθειμένοι. Το μέσο που έχουμε, το Spotlight, το οποίο στόχο είναι να καταπολεμηθεί κάθε είδο βία απέναντι στι γυναίκε και κυρίω ε, ακαταναγκαστική γάμη και ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, αυτό το μέσο λοιπόν πρέπει να ενισχυθεί και να στηριχθεί ευρύτερα από τη διεθνή κοινότητα. Υπάρχει ανάγκη να προβλεφθούν κατά ε, οι ε, δημοσιονομική πόρη για τα ε, δικαιώματα, τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ως προς αυτό βεβαίως θα αντισταθώ στις τροπολογίες που στόχο έχουν να περιορίσουν ή να καταργήσουν τις αναφορές στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Επίσης είδαμε ότι η κοινωνία των πολιτών έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και ιδιαίτερα οι άνδρες και τα αγόρια ε, που έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν στην προώθηση ε, και την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων. Κατά τα λοιπά, βεβαίως εκτίμησα την ποιότητα με πολλών από τις τροπολογίες των συναδέλφων και από αυτής της βάσης είμαι βεβαία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξο και προοδευτικό υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Thank you, Greens. Ευχαριστούμε κυρία Φοφάνα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη δουλειά που κάναμε στην προετοιμασία αυτού του ψηφίσματος και γι' αυτό ο αριθμός των τροπολογιών που υποβλήθηκαν ε, είναι μεγάλος για να μπορέσουμε να έχουμε και πολλές ευκαιρίες να κάνουμε μια δουλειά ε, της προκοπής. Ε, η συνεργασία των Επιτροπών ΔΕΒΕ και ΦΑΜ θα πρέπει να συνεχιστεί για να μπορέσουμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί για τα θέματα αυτά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας πραγματικά ε, μας συγκίνησε ο αριθμός ε, των ε, κοριτσιών και γυναικών σε εγκυμοσύνη και των πόσων προβλημάτων υπήρχαν σε σχέση με την τήρηση των δικαιωμάτων σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας. Η σχολική τους φίτηση είναι πάντοτε μια τροχοπέδη για την ανάπτυξη και πολλές φορές με καταναγκαστικούς γάμους δεν έχουν πρόσβαση στην αναπαραγωγική σεξουαλική υγεία και σοβαρούς φραγμούς για την εξέλιξη αυτών των εφήβων. Είναι μια μορφή βίας γιατί κάθε μέρα μπορούν να δουν τη ζωή τους να καταστρέφεται γιατί κάποιος άλλος αποφάσισε για εκείνες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα τα οποία συζητούμε και να γίνει ένας πραγματικό αγώνας για να φτάσουμε σε επίπεδα μηδενική ενοχής ό,τι αφορά τη βία εις βάρος των γυναικών και κοριτσιών. Επίσης, χαιρετίζουμε την αφοσίωση από τον αγώνα των νέων και θα πρέπει νέοι αυτοί να έχουν κατάλληλη σεξουαλική αγωγή, ε, κατάλληλη για την ηλικία του, που να ανταποκρίνεται στι ανάγκε του, ενώ θα καλύπτουμε και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ισότητα των φίλων προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν ανεξάρτητοι και αυτόνομοι. Επιπλέον θα πρέπει να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις δηλώσεις που κάναμε προφορικά καθώς και τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει να τις επεξεργαστούμε. Χαιρόμαστε λοιπόν για την δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφιερώσει 29 εκατομμύρια ευρώ στην υγεία των νέων και ελπίζουμε ότι το νέο αυτό εργαλείο γειτονία και αναπτυξιακή βοήθεια θα επιτρέψει να, να εκταμιευθούν κονδύλια ώστε να χρηματοδοτήσουμε και άλλε δράσει σε διεθνέ επίπεδο, διότι η αναπαραγωγική υγεία και η χειραφέτηση των γυναικών καθώ και η ισότητα των φύλων είναι ε, παράγοντε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όσον αφορά τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε τα γυναικεία δικαιώματα όπω ε, και τα δικαιώματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι παραβίαση των δικαιωμάτων τη δημοκρατία. Αυτή είναι και μία δήλωση που έχει να κάνει και με τα ε, δικαιώματα που συζητήθηκαν στον Ναϊρόμπι, το δικαίωμα στην αντιψήληψη για παράδειγμα και το πνεύμα τη όλη συνόδου. Θα πρέπει να αποστείλουμε ένα χειρό μήνυμα αλληλεγγύη ε, προ τι γυναίκε και τα κορίτσια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Thank you. Like to one to Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρώμα από το ID. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω και σας και όλους τους συνεργάτες για τη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης. Η σύνοδος στο Ραϊρόμπι ήταν πλούσια σε συναντήσεις, συνομιλίες και σε στοιχεία που πραγματικά μας όκαναν κάποιες φορές. Ε, η μαρτυρία μιας νέας εγγύου, 9, 10 ή 11 ετών, οι κοριτσάκια που έχουν βιαστεί και έχουν καταναγκαστεί σε γάμο, ε, γιατί τις έχει απορρίψει και εκδιώξει η 11 ετων οι κοριτσακια που εχουν βιαστει και εχουν καταναγκαστει σε γαμο γιατι τι εχει απορριψει και εκδιωξει η κοινωνια και η οικογένειά τους. Είναι δύσκολο κανείς ε, να ε, αγνοήσει αυτά τα φαινόμενα ε, και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και πώς. Μέχρι πού πρέπει να πάμε. Με ψηφίσματα, με τροπολογίες και με δωρεές. Θα πρέπει να αποτελέσουμε ένα πρότυπο για να γίνουμε πιο αξιόπιστοι σε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε δει ότι η παραβίαση των γενικών δικαιωμάτων στην Αφρική είναι κάτι το καθημερινό. Τέτοια στοιχεία τα έχουμε λάβει από διαφορετικές μαρτυρίες κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Είναι τεράστιοι αριθμοί που έχουν υποστεί ε, των γυναικών, γυναικείων οργάνων. 41% έχουν ε, καταναγκαστεί σε γάμο πριν τα 18, άλλε τόσε έχουν παντρευτεί πριν τα 18. Η αριθμή αυτή είναι ε, τεράστιε αυτέ τι χώρε. Η παραβίαση των γυναικών δικαιωμάτων στην Αφρική έχει να κάνει και με την ε, ε, εκρηκτική δημογραφική ανάπτυξη που πιέζει και τι θέσει απασχόληση, ε, τα, τα δημοσιονομικά, το κοινωνικό σύστημα και προκαλεί και τεκματικέ αλλαγέ. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτέ τι αναπτυσσόμενε χώρε και να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών. Γι' αυτό έχω αποβάλει σχετικά 17 τροπολογίε από την ομάδα μα. Επιπλέον πρέπει να κοιτάξουμε ότι θα πρέπει να αποτελέσουμε εμεί πρότυπο. Πρέπει να σταματήσουμε να επιτρέπουμε αυτέ τι παραβιάσει γυναικείων δικαιωμάτων να εκδιπλώνονται και στην Ευρώπη. Ε, στη Γαλλία είναι πολλά τα μεγάλη αριθμή των κοριτσιών που έχουν υποστεί ε, ακροτηρισμό των γυναικείων οργάνων. Ε, πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμο σε όλε τι χώρε και κυρίω να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Δεν πρέπει να λυγίσουμε, πρέπει να αντισταθούμε. Σε όλε αυτέ τι πρακτικέ, τι παραδόσει που παραβιάζουν τα γυναικεία δικαιώματα. Πρέπει να δώσουμε παράδειγμα σε όσου αγωνίζονται εδώ στην κλειτοριδεκτομή και να προσπιστούμε τα δικαιώματα των κοριτσιών. Σα ευχαριστώ γιατί η πολύ πλούσια, πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω οι τροπολογίε αυτέ τουλάχιστον μέρη να γίνουν αποδεκτέ. Ευχαριστώ. Thank you so much. Ευχαριστούμε. Και ο λόγος ε, στους σκιώδες εισηγητές των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών της ΓΚΟΥ, αλλά δεν τους βλέπω στην αίθουσα. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να κάνουν σχόλια. Παρακαλώ. Yeah. Any opportunity for... Ναι, οποιαδήποτε ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο, εγώ την παίρνω. Ευχαρίστω. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να συγχαρώ όσους συμμετείχαν στην αποστολή. Ήταν ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Και ξέρω λοιπόν από δική μου πείρα πόσο σημαντική είναι μια τέτοια συμμετοχή. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το ψήφισμα να γίνει όσο το δυνατόν πιο ισχυρό και όπω είπαν πριν και οι συνάδελφοι όσον αφορά την επίθεση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι ταυτόχρονα και επίθεση κατά της δημοκρατίας και το είπαμε και χτε στην ακρόασή μα εδώ στη ΦΑΜ. Έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όλοι είμαστε ίσοι σε αυτόν τον πλανήτη και οι γυναίκε και τα κορίτσια και τα αγόρια. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι ε, θα διασφαλίσουμε οποιαδήποτε δικαίωμα έχουμε αποκτήσει. Δεν θέλουμε να οπισθοχωρήσουμε, να πάμε προς τα πίσω. Και πιο συγκεκριμένα, τα δικαιώματα αυτά αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες. Ε, όλο και περισσότερες επιθέσεις σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε δυναμικά. Δεν έχω τις τροπολογίες, δεν ξέρω αν έχετε αντίγραφα. Απλώς θα ήθελα να σας το αναφέρω. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους για τις δηλώσεις σας και τώρα η Ευλίνα έχει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Θα επαναλάβω αυτά που είπαμε όλοι, ότι οι τροπολογίες αυτές τονίζουν πόσο ξεκάθαρη πρέπει να είναι η διατύπωσή μας επί του θέματος. Να τα πούμε όλα, να είμαστε ισχυροί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις τροπολογίες σας, θα τις λάβουμε υπόψη μας, θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Και όσον αφορά την, το χρονοδιάγραμμα, στις 22 και 23 Ιανουαρίου θα είναι η ψηφοφορία εδώ στη ΦΑΜ. Θα προχωρήσουμε λοιπόν όσο το δυνατό γρηγορότερα για να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Φράνσισα, ήθελα να πω εντάχει ότι θα μπορούσαμε να γράψουμε ε, στην Βουλή της Κένιας για να τους ευχαριστήσουμε για το πρόγραμμα που είχαν δημιουργήσει, γιατί είχαν δεχτεί σημαντική πολιτική πίεση. Ξέρω ότι κάποιες ε, γεγονότα αφαιρέθηκαν από το πρόγραμμα της Βουλής ε, για να δημιουργηθεί το πρόγραμμα και κάποια που έγιναν παράλληλα με την διάσκεψη. Θα θέλαμε λοιπόν να τους γράψουμε για να αναγνωρίσουμε αυτό το πρόγραμμα που κατήρθησαν, που ήταν πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι 150 βουλευτές της Κένια συμμετείχαν. Νομίζω λοιπόν ότι πολιτικά θα ήταν πολύ χρήσιμο να το επισημάνουμε. Εξαίρετη η πρότασή σου. Απλώς πρέπει να σκεφτούμε ποιον θα ευχαριστήσουμε, σε ποιους πρέπει να γράψουμε. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο βεβαίω θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα, διότι πραγματικά η αποστολή ήταν αξιοθαύμαστη. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ατζέντα μας που έχει σχέση με αυτό που αναφέραμε, που είναι η έκθεση της αποστολής μας στο Ναϊρόμπι. Πολλά πράγματα έχουμε ήδη πει, κάποια τα φύξαμε Μαζί με τον Νόμπερτ Νόιζερ, λοιπόν, ε, είχα την ε, τιμή να συμπροεδρεύσω της αποστολής. Ήταν μια πολύ σημαντική αποστολή. Ήμασταν 10 μέλη από την ΦΑΜ και την ΝΤΕΒΕ που συμμετείχαμε στη διάσκεψη κορυφή του Ναϊρόμπι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πήρε το θέμα πολύ σοβαρά και έστειλε ένα δυνατό μήνυμα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω όχι την απλώς καλή, αλλά την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε με την Επιτροπή, το είπε και ο Νόμπερτ Νόιζερ, η ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήθελε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αυτή ήταν η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακούστηκε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιοι αναφέρατε ήδη τη συνέντευξη τύπου και το μήνυμα που στείλαμε λοιπόν στο κοινό. Συναντηθήκαμε με μη κυβερνητικέ οργανώσει, πολύ σημαντικές. Δώσατε κάποια σημαντικά παραδείγματα, όπως το Deutsche Stiftung και άλλε τοπικέ ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει. Συναντηθήκαμε με γυναίκε από την Κένια και ε, επίσης ε, το, ένα, μια εκπομπή να ε, τηλε-reality show το οποίο χρηματοδοτούμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κένια. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι αυτή η αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να συμμετέχει με την ίδια προθυμία και στο μέλλον για την ε, διασπορά της γνώσης, της εμπειρογνωμοσύνης, για να συμμετέχουμε πιο ενεργά σε ε, διεθνείς ε, διασκέψεις κορυφές, κορυφής. Διότι εκεί ακριβώς έχουμε την ευκαιρία να εντείνουμε, να κάνουμε σημαντικότερες τις διεθνείς μας σχέσεις. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι συμμετείχαμε και στις ε, διαφορετικές συνεδριάσεις διασκέψης κορυφής, αλλά και το φόρουμ που έγινε ε, με τη ε, συμμετοχή των μελών της Βουλής για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Υπήρχαν σημαντικά πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε εκεί και βεβαίως θα θέλαμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση μας. Συναντήσαμε επίσης την Νατάλια Κανέμ, ε, εκτελεστική διευθύντρια του UNFPA, που ήταν και η κινητήριος ε, δύναμη για όλη αυτή τη διάσκεψη κορυφής. Και για να κάνουμε μια περίληψη, αν κατακλείδει, μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε το ρόλο που εμείς ως ε, Ευρωκοινοβούλιο μπορούμε να παίξουμε σε αυτό το διεθνές πεδίο. Οπωσδήποτε, το είπαμε και στην συνέντευξη τύπου, πριν αυτή τον είπα και μετά από αυτή της Αγίας Έδρας, ότι είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο, ότι τα δικαιώματα των γυναικών, η δημοκρατία, η εκπαίδευση, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ότι αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας και εγώ ως συμπροεδρεύουσα λοιπόν της αποστολής θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη της αποστολής που πραγματικά εργάστηκαν στενά και με αγαστό πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα του Ευρωκοινοβουλίου και βεβαίως ε, το ίδιο θα κάνουμε και σε μελλοντικές εκδηλώσεις ε, τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως ε, θα συνεργαστούμε στενά και με την ΤΕΒΕ. Αυτά και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Όμπερτ Νόιζερ που έχει ήδη κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια για να μας δώσει την άποψη της ΔΕΒΕ αλλά και στους συμμετέχοντες στην αποστολή ίσως. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Να τον πάρει και πάλι ή όχι. Πιερέτ. Να επαναλάβω ότι ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία Απλώς κάτι που προσωπικά με εντυπωσίασε ήταν η συμμετοχή, ε, κυρίως η αφοσίωση και το πάθος των νέων. Αυτό για μένα ήταν κάτι καινούριο. Έχω πάρει μέρος σε πολλές διασκέψεις, στο Πεκίνο ας πούμε. Ε, οι νέοι ε, αποκλείονταν ουσιαστικά, δεν μπορούσαν να έχουν συμμετοχή. Αυτή τη φορά πραγματικά είχαμε την εντύπωση ότι εκείνοι θέλουν να αναλάβουν την, αλλαγή που, την ευθύνη για την αλλαγή που πρέπει να γίνει στη σεξουαλική αγωγή. Και δεν θα έλεγα ότι είναι πολιτική κάποια συγκεκριμένη χώρα, αλλά κάποιων αφρικανικών χωρών να αρνούνται την πρόσβαση στην σεξουαλική αγωγή. Θα πρέπει, ενώ άλλες το ζητούν, ε, το ζητούν επίμονα. Θα πρέπει λοιπόν, ήσασταν εκεί. Ε, Μα είπαν οι νέοι ότι δεν θέλουμε να, να γίνεται πια αυτό, δεν θέλουμε να βιάζονται τα κορίτσια, δεν θέλουμε να τι υποχρώνουν να παντρεύονται έτσι. Τι να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτό. Και όλοι τόνισαν ότι η σεξουαλική αγωγή πολλές φορές ε, επικεντρώνεται στον οικογενειακό σχεδιασμό. Δεν χρειάζονται αυτό μόνο. Ε, θέλουν τη θέση τους ε, και διεκδίκησαν τη θέση τους αυτό το φόρουμ. Μάλιστα πρόβαλαν πολύ έντονα τις επιθυμίες τους, αυτά που θέλουν για να φτάσει επιτέλους η στιγμή της αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης. άλλος κανείς, τότε απλώς να πω ότι ε, συμφωνώ απολύτως με αυτό που μόλις είπατε. Πραγματικά η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός νέων ανδρών και γυναικών, νέων ανθρώπων, με όλες τους τις προσπάθειες, πραγματικά ενισχύουν την αξιοπιστία όλων αυτών που γίνονται. Διότι όταν οι νέοι έρχονται σε επαφή με μας και αγωνίζονται δικαιώματα, Φυσικά ε, η αξιοπιστία μας ενισχύεται και αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εάν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μιλτάντα, Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, για να μας πει τις απόψεις του για τα ε, συμπεράσματα της Συνόδου. Α, εδώ είστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη εισαγωγή για το EPF και το ρόλο στην ε, διάσκεψη. Για το τι κάναμε εμείς στο Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα. εμείς ασχοληθήκαμε ως Διευθύνουσα Επιτροπή μαζί με την κυβέρνηση της Κένια και το Φάντα ε, του ΟΗΕ για τα θέματα αυτά και το φόρουμ των βουλευτών που γινόταν παράλληλα ε, με την Σύνοδο. Τρία πράγματα θέλω να πω σε σχέση με τη δουλειά του Ευρωκοινοβουλίου εδώ και τη Σύνοδο. Πρώτον, Θέλω να συγχαρώ την αντιπροσωπεία και την πρωτοβουλία των Επιτροπών ΦΑΜ και ΝΤΕΒΕ να πάρουν μέρος με τόσο έντονο τρόπο στην ε, σύνοδο αυτή. Ήσασταν πραγματικά μεταξύ των τριών μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών που πήραν μέρος μαζί με αυτή τη βουλή τη Κένια βεβαίω και τη Δανία. Η παρουσία της Ευρώπης ήταν πολύ σημαντική, σημειώθηκε και έγινε αισθητή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ, όταν μιλάμε για αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα που ξέρουμε ότι απειλούνται ε, το ακούσαμε από πολλούς συναδέλφους σας εδώ και το έχουμε ακούσει και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, οι αμφιβολίες για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών που έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει σημειωθεί και είναι και κάτι για το οποίο πολλοί λυπούνται. Όμως, ακούσαμε από διαφορετικές πλευρές ότι υπάρχει διπλωματική πίεση από τη ΣΥΠΑ σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο, σε διαφορετικές χώρες, να μην προσυπογράψουν τη δήλωση του Ναϊρόμπι. Και αυτό πραγματικά έχει πετύχει σε μια χούφτα περιπτώσεων, Όλο λοιπόν που είναι κάτι το οποίο δυσαρεστεί, έχει δυστυχώς ε, θεωρηθεί ένα βήμα αποτυχίας. Και τώρα για την καθολικότητα της δήλωσης του Ναϊρόμπι και το πρόγραμμα δράσης για τα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπολικής υγείας. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα δράσης για χώρες που αφορά το νότο του υδρογείου ή τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι κάτι που αφορά και τις χώρες μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον οικογενειακό σχεδιασμό πολλά μπορούν να γίνουν για την πρόσβαση σε αυτόν και στην Ευρώπη, αλλά και ε, στο Νότο και για την ε, υγεία. Ακούσαμε και για την Ευρώπη, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μετανάστες, Ρωμά και ούτω καθεξής. Ε, εδώ επίσης μας ενδιαφέρει και η πρόσβαση στην αντισύλληψη ε, πρέπει να ασχοληθούμε με τα δικαιώματα της προστασίας αυτής, ε, τα δικαι... την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί και σίγουρα υπάρχουν ε, τέτοιες επιζήμιες πρακτικές στο νόδο της Ιδρογείου, Global South και πλήττονται κυρίως γυναίκες και κορίτσια. Ε, όλες αυτές οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες, αλλά έχουν γίνει και έρευνες ώστε να τιμολογήσουμε την ε, χρηματική, την οικονομική αξία τη κάθε προσπάθεια και να δούμε πώ μπορεί να πετύχουμε και με πόσα κονδύλια βελτίωση στην κάθε περίπτωση. 264 δις δολάρια χρειάστηκαν την τελευταία δεκαετία για τέτοιου αριθμού. Είναι ένα ε, αριθμό εντυπωσιακό, αλλά σίγουρα απαραίτητο. Και η δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 29 εκατομμύρια για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι ευπρόσδεκτη. Και μετά, τελευταία παρατήρηση για τι τροπολογίε που έχουν αποβληθεί για το ψήφισμα αυτό. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο να είναι αποτελεσματικό. Επειδή υπάρχει ε, διαφωνία απόψεων εδώ, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην θεωρηθεί μόνο μια πηγή χρηματοδότηση για την και βοήθεια, αλλά πραγματικά και ένα θεματοφύλακα των ε, καθολικών αξιών, των οικουμενικών αξιών. Ας πούμε, στις τροπολογίες λοιπόν, καλό θα ήταν να γίνει αναφορά και στις αναθεωρήσεις του ICPD που έγιναν μετά από το φόρουμ και επίσης να αναφερθούμε και στην διάσκεψη ΕΨΗ, την Διεθνή Διάσκεψη των Βουλευτών, την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη, γιατί σε πολλές χώρες είναι μια από τις βασικές πηγές για να ξεκινήσουν κάποια βήματα πρόοδου σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, έγινε αναφορά ε, στην, ε, στην περιοριστική θεώρηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των μητέρων, των μητέρων και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Θα πρέπει αυτό να αλλάξει, καθώς θα πρέπει και οι επίτροποι Γιουπιλάιναν και Ντάλι να αναλάβουν, ε, να φέρουν εις πέρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much and uh, also for the way of cooperation. Σας ευχαριστώ πολύ και για το τρόπο συνεργασίας που πραγματικά ε, ήταν κάτι που πραγματικά μας ε, εμπλούτησε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Φρανθίσκο, Φρανθίσκο Λόπες. Παρακαλώ. Είμαι ο Φρανσίσκο Γκαρσία. Δυστυχώς η Ανδριέτ Γκέγκερ, η διευθύντριά μου, δεν, ήταν, ε, δεν μπόρεσε να είναι εδώ στην ώρα της γιατί ήταν σε, ε, αναγκάστηκε να είναι σε μια άλλη συνεδρία. σε ξενόματός της θα ήθελα να συγχαρώ ε, και τις δύο επιτροπές για την παρουσία σας στον Αϊρόμπ. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό και η διευθύντριά μας ήταν επίσης πολύ ικανοποιημένη και υπογράμμισε και την εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο πράγμα που οδήγησε σε πραγματικά ισχυρή παρουσία της Ένωσης στο Ναϊρόμπι και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο για τη στήριξη των γενικών δικαιωμάτων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διευθυντριά μου συμμετείχε σε τέσσερα πάνελ και ήταν πολύ ευχαριστημένη που μπόρεσε να ανακοινώσει 29 εκατομμύρια σε αυτή τη διαδικασία και επίσης νέες δεσμεύσεις ανακοίνωσε για 100 εκατομμύρια για αυτή την ε, πρωτοβουλία Spotlight ε, για την καταπολέμηση της βίας. Είδαμε ε, από την έκθεση της, της αποστολής την ότι εγκρίνουμε όλοι και συστήνουμε τη συνεργασία. Ε, το θέμα βέβαια είναι τώρα να δώσουμε συνέχεια σε όλα αυτά. Εμείς είμαστε πάντως πανέτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και να δουλέψουμε για αυτές μας τις ε, ε, δεσμεύσεις. Πρόεδρος, προσβλέπουμε και εμείς την συνεργασία και τώρα με αυτές τις παρατηρήσεις, το σχέδιο της αναφοράς για την αποστολή είναι στους φακέλους σας και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση λοιπόν, οπότε εγκρίνεται και δίνω το λόγο τώρα στο Συμπρόεδρο. Ναι. Θα ήθελα και εγώ άλλη μια φορά να ευχαριστήσω του συμπροέδρους της αποστολής και φυσικά όλα τα μέλη που έκαναν πολύ σημαντικό έργο. Πιστεύω πως μετά από αυτή την κοινή αποστολή και σας διαβεβαιώ ότι και από πλευράς ΔΕΒΕ θα κάνουμε το αίτημα για να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να δράσουμε από κοινού όταν θα γίνει τον επόμενο χρόνο η διάσκεψη για τις γυναίκες στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Εμείς Είμαστε στην ώρα μας, έχουμε δύο λεπτά. Δεν θέλω να κάνω διάλειμμα, αλλά θέλω να περάσω κατευθείαν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας μας διάταξη που θα συνεχίσει τη συνεδρίαση μόνο η δική μας Επιτροπή, Επιτροπή ΦΑΜ. Ευχαριστώ πολύ σε, όλους, σε όλα τα μέλη της ΔΕΒΕ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.